συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. Θα δώσουμε καταρχήν το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ρενάτο Σόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας ε, με το οποίο ασχολήθηκα το τελευταίο 1,5 χρόνο ε, και που ελπίζω ότι αύριο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς ε, με την ψηφοφορία. Πρόκειται ακριβώς για την Security Financing Transaction όπως είναι ο τίτλος στα αγγλικά και που σημαίνει διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. Με μεγάλη χαρά δούλεψα για το θέμα αυτό ε, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά και γιατί θεωρώ ότι επιτύχαμε ε, τους ε, δύο κύριους στόχους, δηλαδή να διασφαλίσουμε αγορά με ρευστότητα για τις συναλλαγές μεσοτήτρων, αλλά κυρίως να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και καθαρούς κανόνες με τρόπο ώστε να αποφευθούν οι συστημικοί κίνδυνοι της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Η κρίση του 2007 στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, που με πολύ έντονο τρόπο μετατοπίστηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, για, ε, απέδειξε ότι το τραπεζικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διασυνδεδεμένο. Επίσης και ότι είναι πάρα πολλές διασυνδέσεις ανάμεσα στην παραδοσιακή τραπεζική αγορά ε, και την λεγόμενη σκιώδη ε, τραπεζική ε, αγορά. Και υπάρχουν πάρα πολλές συναλλαγές οι οποίες γίνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός όμως του πλαισίου εντός του οποίου οφείλουν να κινούνται. Η Κεντρική Τράπεζα είπε κάποια στιγμή ότι το σύστημα του shadow banking είναι πάρα πολύ μεγάλο, υπερβολικά μεγάλο και υπερβολικά ε, χρεωμένο. Ε, αυτός ακριβώς ο υπερβολικός βαθμός ε, χρέωσης αύξησε τον κίνδυνο αλλά και την επικινδυνότητα του συστήματος στο σύνολό του. Το shadow banking μπορεί να εκπροσωπεί το 2011 περίπου δολάρια, δηλαδή, ευρώ, συγγνώμη, δηλαδή τέσσερις φορές το συνολικό ΑΕΠ της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση μέσω ε, τίτλων αποτελεί ένα σημαντικό ένα ε, σημαντικό στοιχείο διασύνδεσης ανάμεσα στην παραδοσιακή τραπεζική αγορά και το σκιώδες ε, τραπεζικό ε, σύστημα. Η ομάδα υψηλού επίπεδου υπό τον Λικάνεν στην αρχή και υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά δούλεψε έτσι ώστε να διασφαλίσει ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί με νόμους διαφάνειας και πιστότητα, αλλά που ε, δεν θα εμποδίζει την ρευστότητα και την χρήση τη ρευστότητα αυτής. Ο κανονισμός που θα ε, κληθούμε να εγκρίνουμε ε, στοχεύει να βελτιώσει τρία συγκεκριμένα στοιχεία αυτής της αγοράς. Πρώτα απ' όλα ο κανονισμός που προτείνεται προτείνει όλες ε, οι ε, συναλλαγές ε, να καταγράφονται σε ένα κεντρικό database, σε μια κεντρική τράπεζα δεδομένων, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιε είναι ακριβώ οι διασυνδέσει και του τραπεζικού συστήματο και παραδοσιακού τραπεζικού συστήματο. Δεύτερον, διαφάνεια ανάμεσα στους επενδυτικούς, στα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία επενδύονται και τους επενδυτές και τέλος καλύτερη ρύθμιση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποίησης ε, των ε, τίτλων επανυποθήκευση δηλαδή των βεβαίω μπορούν εδώ να συντείνουν και να ε, χρησιμοποιηθούν και άλλες ρυθμίσεις ε, όπως ε, ας πούμε το ΕΜΙΡ που αφορούν ακριβώς τον ίδιο τομέα. Είναι σημαντικό να συνδυάσουμε την διαφάνεια μαζί με την ασφάλεια των συναλλαγών και αυτό υπό την εποπτεία και της Κεντρικής Τράπεζας. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα καλό συμβιβασμό ο οποίος θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια αύριο. Ε, ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν, τον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα την ευκαιρία να συζητήσω τον κανονισμό για τις ε, συναλλαγές σε αξιόγραφα και ευχαριστώ τον κύριο Σόρου και τους σκιώδεις συγητές του για το έργο το οποίο έχουν φέρει σε πέρας. Αυτός ο κανονισμός είναι τμήμα της απάντησής μας για τα προβλήματα που υπήρξαν στις χρηματαγορές θα δημιουργήσει περισσότερη ασφάλεια, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην ε, σκιώδη τραπεζική ε, δραστηριότητα και να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020 συνοδεύει άλλα μέτρα που έχουμε ήδη λάβει για να τυθασεύσουμε τον τομέα της σκιώδους τραπεζικής ε, δράσης. Ε, οι χάρη, προηγούμενοι κανονισμοί για τις εναλλακτικέ επενδύσεις και τα παράγωγα ρυθμίσουν τις αγορές αυτές. Όλοι αυτοί που παρακολούθησαν αυτή την ε, έκθεση ξέρουν ότι οι συναλλαγές ε, όπου χρησιμοποιούνται ως έγκυα τα αξιόγραφα είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις χρηματαγορές της Ευρώπης. Υποστηρίζουν τις επενδύσεις και επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Κατά τη διάρκεια τη κρίση, τη χρηματοπιστωτική κρίση, ήταν σαφέ ότι δεν ξέραμε αρκετά για το τι γίνεται σε αυτέ τι αγορέ. Χωρί αξιόπιστα στοιχεία δεν μπορούμε να ξέρουμε αρκετά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συστημικού κινδύνου τόνισε ότι με μεγαλύτερη διαφάνεια θα ξέρουμε καλύτερα ποιο είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και θα μπορούμε να τους ελέγχουμε και να παίρνουμε καλύτερε επενδυτικέ αποφάσει. Αυτή ήταν και η ανάλυση Κομισιόν. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που είμαστε πολύ κοντά στο να φτάσουμε μια τελική <clears throat> συμφωνία για μια νομοθεσία η οποία θα αυξήσει τη διαφάνεια. Είμαι ευγνώμων για το Κοινοβούλιο για το καταπληκτικό αυτό έργο που έχει κάνει και πιστεύω ότι και στην συνεννόηση με το Συμβουλίο θα πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε τις ε, αναφορές σε των ε, συναλλαγών σε κεντρικά αποθετήρια συναλλαγών σε τράπεζες δεδομένων όπου μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δεύτερον, θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους επενδυτές, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ε, εκθέσεις για τα αξιόγραφα, αλλά και για τις προτάσεις πριν από τις επενδύσεις, ώστε να μπορούν να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Τρίτον, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για την επαναχρησιμοποίηση των αξιογράφων ως εχεγείων. Γιατί έτσι μπορούν να αποφευθούν φαινόμενα ντόμινο όπως αυτά τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση των βορείων βράχων, της Northern Rocks δηλαδή. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη υποδομή στις χρηματαγορές. Με ένα πίνακα λοιπόν ε, για όλες αυτές τις συναλλαγές θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έτσι θα μειωθεί και το βάρο στι μικρομεσαίας επιχειρήσει και θα διατηρηθούν μονάχα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για αριθμιστικού και εποπτικού σκόπου. Ο αριθμό των αριθμιστών που μπορούν να ε, έχουν πρόσβαση σε αυτά έχει τροποποιηθεί για να υπάρχει συνεκτικότητα σε όλα αυτά. Η αρχή αγορών αξιογράφων θα δημιουργήσει και τις απαραίτητες ρήτρε για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Η ΕΣΜΑ θα εξασφαλίσει λοιπόν μια ισόρροπη εφαρμογή σε όλε τι χρηματαγορές. Η Κομισιόν παραμένει στα πλαίσια μια σωστή ισορροπία με αναλογική ρύθμιση ώστε να διατηρηθεί και η διαφάνεια αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη ατζέντα. Με το να υπάρχουν όλε αυτέ τι πληροφορίε, μπορούμε να βοηθήσουμε του επενδυτέ να έχουν τι κατάλληλε αποφάσεις και να έχουν μια ε, υπεύθυνη στάση, να αποφύγουμε τις κρίσεις και να μπορούμε να παρέμβουμε όταν χρειάζεται από στοιχείων ο κανονισμός για τις συναλλαγές αξιογράφων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Προσβλέπω στην επερχόμενη συζήτηση και την ψήφιση της έκθεσης αύριο, την Πέμπτη δηλαδή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων εκ μέρους του ΕΛΚ. Η κυρία Ντανούτα Μαρία Χιούμπνερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Ντομπρόσκη, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο νέος ε, κανονισμός ε, θα φέρει άλλο ένα βαθμό διαφάνειας ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ποιος συναλλάσσεται με ποιον και υπό ποιες συνθήκες. Αυτό θα βοηθήσει τους φορείς της αγοράς. Επίσης, η διαφάνεια μπορεί να εμποδίσει την μετακίνηση συναλλαγών από το τραπεζικό σύστημα στο λιγότερο ρυθμισμένο ε, σύστημα εκτός των τραπεζικών συναλλαγών. Επίσης, η ΟΣΕΚΑ και ε, το σύστημα ενημέρωσης των επενδυτών θα βελτιωθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό αυτό για να γίνουν δύο τροπολογίες στον κανονισμό ΕΜΙΡ. Να έχουμε πρόσβαση τις πληροφορίες που υπάρχουν στα αρχεία καταγραφής ε, συναλλαγών, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι αρχές εξυγίανσης να έχουν καλή πρόσβαση στα στοιχεία της εποπτείας. Θα είναι πιο εύκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βλέπει τις ρυθμίσεις ε, τρίτων χωρών και να βλέπει αν είναι ισοδύναμες με αυτά τα οποία απαιτεί ο κανονισμός ΕΜΙΡ. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρούνται από κάποιες ε, ε, υποχρεώσεις γιατί ο αντισυμβαλόμενος θα πρέπει να υποβάλει την έκθεση εκ μέρους και των δύο συμβαλωμένων σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, κ. Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή, τον Ρενάτο Σόρου, για το έργο αυτό που έφερε πέρασε εδώ και δύο μήνε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Ολομέλη και να γίνει αύριο η ψηφοφορία του κανονισμού αυτού. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την αδιαφάνεια που υπάρχει και τις συμφωνίες εκτός ρυθμισμένων αγορών σε ό,τι αφορά πωλήσει αξιογράφων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε νέες λειτουργίες στο σύστημα ανάλυσης και εποπτείας των χρηματαγορών και να υπάρξει καλύτερη ροή πληροφοριών για όλους τους παίκτες στον χώρο της αγοράς. Νομίζω λοιπόν ότι επέτυχε ο κύριο Σόρου μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση ότι μέσα σε αυτό το πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την Ένωση Κέφαλη Αγορών θέλουμε αυτή η Ένωση Κέφαλη Αγορών να μην οδηγήσει σε νέους τρόπους που να εκφεύγουν του ελέγχου μέσω του shadow banking, της σκιώδους τραπεζικής δραστηριότητας. Θέλουμε να έχουμε μια διάφανη και εποπτευόμενη τραπεζική λειτουργία και λειτουργία αξιογράφων, μόνο επί αυτή τη βάση μπορούμε να φτιάξουμε την Ένωση Κεφαλαίου Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Από την ομάδα του ECR, ο κ. Όζοκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο πρώτος στόχος της έκθεσης αυτής είναι να αυξήσει την ε, οικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί εάν βελτιώσουμε τη διαφάνεια αυτών των συναλλαγών. τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και άλλες δραστηριότητες αντίστοιχες. Η πολιτική ομάδα του ECR στη συνεργασία με το ΕΛΚ και με τους φιλελεύθερους ε, θα υποβάλουν τροπολογίες και χάρη στις τροπολογίες αυτές πιστεύουμε ότι ε, διευκρινίζουμε κάποιες αμφιβολίες που υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη μειώνουμε τις ε, προϋποθέσεις σε σχέση με την υποβολή πληροφοριών για τις εισηγμένες εταιρείε. Επίσης, ε, και όσον αφορά την ε, διάταξη σχετικά με την παροχή εγγύησεων. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων, Φιλίπ Τεμπάκερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ενδεχομένως δεν είναι η πιο έντονη συζήτηση που θα ακούσει κανείς σήμερα στο Κοινοβούλιο, σήμερα το βράδυ. Ωστόσο πιστεύω ότι ολοκληρώνοντας τη συζήτηση αυτή ε, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι ε, συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο τμήμα των συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το καλό όλων των συναλλασσομένων αλλά και για την επίτευξη χρηματοπιστωτική σταθερότητας. Και επομένως ε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ε, με τον σωστό τρόπο ε, ε, σημαντικά βήματα ε, γίνονται σε τρεις τομείς. Πρώτον όσον αφορά το reporting επίσης με τον τρόπο αυτό μειώνεται το βάρος των μη χρηματοδοτικών εταίρων ας πούμε της μικρομεσαίας επιρρήχησης. Δεύτερον διασφαλίζεται η διαφάνεια προς τους επενδυτές. Τα funds πρέπει είναι υποχρεωμένα πλέον να κοινοποιούν ακόμα και τους κινδύνους ως πούμε των επενδυτικών μέτρων τους. Επίσης, ε, ε, ε, η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, η επαναπόληση τίτλων. Οι τίτλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονάχα υπό συγκεκριμένε παραμέτρους και μονάχα σε περίπτωση κατά την οποία δεν αφορά Ε, Επίσης το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη τα οποία είδαμε στην ελοπίση του ΕΜΙΡ και να αποφύγουμε ε, αποκλεισμούς και αδιέξοδα. Θα πρέπει όλες οι χώρες να ε, υλοποιήσουν στο βαθμό που πρέπει ε, το δικό το κομμάτι που τους αρμόζει. Με τον τρόπο αυτό και ολοκληρώνω θα πρέπει να θα δημιουργήσουμε μια τραπεζική αγορά με ελάχιστο βάρος και άχθος για όλους και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσετε όλοι την υπερψήφιση της Εκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπερνάρ μόνο για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, η παράλληλη αγορά, η σκιώδης τραπεζική αγορά αφορά, ε, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας. Η χρήση τοξικών εργαλείων ε, χειροτερεύει ακόμα την κατάσταση. 3 εκατομμύρια δολάρια εκτός ισολογισμού κυκλοφορούν στην τραπεζική ελληνική αγορά ε, και επομένως είναι σημαντικό και για τις ε, αγορές αλλά και για τις ε, εισηγμένες επιχειρήσεις να υπάρχει διαφάνεια αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δημόσιες συναλλαγές καθώς επίσης και οι συναλλαγές που αφορούν την επαναπόληση. Οι τράπεζες, οι παραδοσιακές, οι οποίες χρησιμοποιούν για τις επενδύσεις, τις αποταμιεύσεις και τις καταθέσεις ε, δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να συνεχιστεί. Ε, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα χρήματα των αποταμιευτών δημοσίων ή ιδιωτικών έτσι ώστε να σωθούν οι αποτυχημένε, ε, εφαλειρημένε τράπεζες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόμτς, μισή λεπτό. Ευχαριστώ Η παγκόσμια κρίση μεταξύ άλλων μας έδειξε πολλά σφάλματα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Μας έδειξε πώς πολύ γρήγορα μπορούμε να φτάσουμε και σε εγκληματικές ακόμη ενέργειες που οδηγούν σε τεράστια κέρδη. Παράλληλα με το γρήγορο κέρδος, συχνά έρχονται και οι μεγάλες απώλειες. Θέλουμε να εμποδίσουμε, θέλουμε να αποτρέψουμε το να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι και οι καταθέτες από αυτά τα σφάλματα. Θέλω να αναφέρω το εξής. Στην Σλοβενία έχουμε μεγάλα προβλήματα με τον τραπεζικό τομέα έχουν επιβαρυνθεί σε μεγάλο βαθμό οι φορολογούμενοι και ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Όταν το κόμμα μας στην Σλοβενία ζήτησε να μάθει τι ακριβώς συνέβη στον τραπεζικό τομέα, πάντοτε μας έδιναν την ίδια απάντηση, ότι αυτά είναι τραπεζικό απόρριτο. Και βέβαια είναι σημαντικό το τραπεζικό απόρριτο, αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι συνεχώς θα εκμεταλλεύονται αυτή την αρχή και δεν θα μας δίνουν απαντήσεις. Θα πρέπει και στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύσουν αυτοί οι κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νίνα Γκίλ έχει το λόγο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίστροπε. Συγχαρητήρια στο Ρενάτο όλο τον καλό μου συνάδελφο, για μια θαυμάσια έκθεση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι στο μέλλον θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, συναλλαγές αξιογράφων ο στόχος των αναφορών σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές είναι να υπάρξει μεγαλύτερη εποπτεία και καλύτερη διαφάνεια. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές αυτές αξιογράφων οι οποίες δημιουργούν ρευστότητα και εξασφαλίζουν καλύτερη χρησιμοποίηση κεφαλαιοϊκών πόρων και έτσι ενισχύονται όχι μονάχα υποχρεώσεις παροχής αναφορών υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που επιτρέπουν την καλύτερη ε, εποπτεία του, της συγκέντρωσης του κύκλου, του, του κινδύνου και έτσι ευνοούν <clears throat> τις αγορές. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε μονάχα να έχουμε ρυθμίσει στον τραπεζικό τομέα. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε και όλες τις άλλες δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο σκιώδη τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ρόλο έχει η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση είναι φανερό ότι ο έλεγχο δεν πρέπει να βελτιωθεί μόνο στον παραδοσιακό ε, τραπεζικό τομέα αλλά και στις τράπεζες επενδύσεων. Ο η δραστηριότητα των τραπεζών έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα παρά το γεγονός ότι είναι μια ανθούσα χρηματοπιστική δραστηριότητα. Όπως τονίζεται λοιπόν από την ε, έκθεση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι συναλλαγές αξιογράφων βοηθούν με την καλύτερη κατανομή των επενδύσεων, αλλά μπορούν να δώσουν δυνατότητα δημιουργία φυσαλίδων με την σκιώδη τραπεζική ε, δραστηριότητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει απαραίτητη εποπτεία και διαφάνεια, ώστε θα πρέπει να είναι σαφές πότε εμπλέκονται σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στα χρηματιστήρια. Με τη νέα αυτή διαφάνεια θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένα τα το κόστος που θα επομιστούν οι νέες οι επιχειρήσεις και πρέπει να ρυθμιστούν όλες οι εκτός ρυθμισμένων αγορών στις συναλλαγές over the counter. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο επιτυχάνει η έκταση και γι' αυτό θα ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μαν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαφώς έχει κάνει πρόοδους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποπτεία και η ρύθμιση θα πρέπει να βελτιωθούν όχι μόνο στον τραπεζικό τομέα αλλά και στον μη τραπεζικό τομέα και θα πρέπει να ρίξουμε φως και στον μη τραπεζικό τομέα στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί και να αποτρέπει τους ε, πιθανούς κινδύνους και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση. Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να υπάρξουν σημαντικές παρενέργειες μόχλευσης. Η συνάδελφος ε, Ντανούτα Χιουμπνέρ από το ΕΛΚ έχει δίκιο όταν ε, ανέφερε ε, ότι οι επιπλέον ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεταφορά των δραστηριοτήτων από το τραπεζικό σύστημα στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Χρειάζονται σαφείς ρυθμίσεις και σαφείς κυρώσεις. Χαίρομαι ε, για τις ε, ε, συζητήσεις που γίνονται και στον τριμερή διάλογο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε να έχουμε σημαντική πρόοδο και διαφάνεια. Συμφωνώ λοιπόν με την Επιτροπή γι' αυτό. Οι συναλλαγές χρηματοδότηση τίτλων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να αποφεύγεται και η επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να παραμένει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κύριε Σάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε τράπεζε και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που να λειτουργούν με βάση διαφανεί κανονισμού. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει και αποπληθωρισμός. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κενό επενδύσεων και η διαφάνεια δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια περαιτέρω κρίση του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ όλων των θεμάτων που μας ενδιαφέρει. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά που κάνουμε για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων ε, θα ε, συμβαδίζουν με αυτά τα οποία απαιτεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει μηνύματα διφορούμενα από τη μια μεριά να λέει στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ε, δράσουν ενεργά από την άλλη μεριά να τους εμποδίζει στις συναλλαγές τους. Θα πρέπει ε, αυτά τα οποία κάνουμε να αποτρέπουν ε, τους υψηλούς κινδύνους για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Αλέθια Μαρία Μόσκα. Ένα λεπτό. Από ό,τι βλέπω απουσιάζει. Δεν πειράζει. Ξεκινάει η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Στάνισλαφ Πόλτσακ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι θα πρέπει να ρίξουμε περισσότερο φως ε, σε αυτήν την σκοτεινή σκιώδη τραπεζική αγορά όπου φαίνεται να λειτουργούν ανενόχλητες μέχρι τώρα οι τράπεζες. Ένας από τους συναδέλφους εδώ είπε ότι ο διαχωρισμός των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων των τραπεζών από τις άλλες δραστηριότητες ε, είναι ένας τρόπος. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτός ο τρόπος, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στις τραπεζικές δραστηριότητες και με αυτό συμφωνούμε όλοι θα πρέπει να σταματήσουν οι υψηλά, υψηλού κινδύνου και κερδοσκοπικές δραστηριότητες ε, που έχουν και πολλά, πολλές παράπλευρες ε, απώλειες και εν πάση περιπτώσει οδήγησαν ε, και στην κρίση την οποία είδαμε τα τελευταία χρόνια. Ε, επίσης, ε, μέσω της προτάσεως γίνεται προσπάθεια να μειωθεί ε, το διοικητικό άκθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό μας ικανοποιεί απολύτως. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σάνι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι ότι ο κίνδυνος ε, είναι μεγάλος όσον αφορά ε, τον τραπεζικό ε, σκιώδη τομέα. Αυτό το είχε, είχε καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό ξεκίνησε τις διαδικασίες έτσι ώστε να σταματήσει πλέον αυτή η διαφανής δραστηριότητα. Τώρα γνωρίζουμε καλύτερα το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ωστόσο αυτό το σύστημα, το παράδειγμα παράλληλο τραπεζικό σύστημα ε, έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από ε, τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει από το ρυθμό αντίδρασης ε, της Ευρώπης. Να πω λοιπόν στην Κομισιόν ότι θα πρέπει με ταχύτητα να προχωρήσει στο δρόμο που έχει καθορίσει και εμείς θα την στηρίξουμε οι προκλήσεις ε, είναι ε, σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει, πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγάλη ταχύτητα αυτόν τον γοργά αναπτυσσόμενο ε, σκιώδη τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα σε αναπληρώτης Νότης Μαριάς. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η τραπεζική κρίση του 2008 και η φούσκα των στεγαστικών δανείων και των subprimes έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη για διαφάνεια στη συναλλαγή τίτλων προκειμένου να υπάρξει ισορροπία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αποφευχθούν στο μέλλον νέε κρίσει. και διαφάνεια σημαίνει αναλυτικέ αναφορέ σχετικά με τι εξασφαλίσει που υπάρχουν για του διάφορου τίτλου. διαφάνεια σημαίνει υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να γνωστοποιούν στου αγοραστέ τίτλων όλους τους πιθανούς κινδύνους. διαφάνεια σημαίνει έλεγχο στο λεγόμενο σκιώδες τραπεζικό σύστημα που αναπτύσσεται με ηλικιώδη ταχύτητα και δημιουργεί υπερβολική μόχλευση κεφαλαίων. διαφάνεια σημαίνει να γνωρίζει η ίδια η κοινωνία πού κατευθύνονται τα κεφάλαια κατευθύνονται στη χρηματοδότηση της παραγωγικής οικονομίας ή στην κερδοσκοπία διότι για να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση πρέπει να μπει τέλος στην οικονομία καζίνο. ευχαριστώ. Μάρκο Βάλι. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σκιώδες τραπεζικό σύστημα είναι αυτό ε, το οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο τμήμα του συστημικού κινδύνου και εν μέρη ε, ε, εν σε αυτό οφείλεται η μεγάλη κρίση. Η χρήση τώρα των οι συναλλαγές αγοράς επαναπόλησης καθώς επίσης και το θέμα των εχεγγύων είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς όμως οι δύο τελευταίες διατάξεις Banking Reform καθώς επίσης και αυτό το οποίο μας απασχολεί σήμερα είναι περιορισμένα, έλειψε η σημαντική πολιτική βούληση γιατί στην ουσία εμείς θέλουμε Capital Market Union και δυνατότητα ε, χρήσης και επαναχρήσης ε, παραδοσιακών ε, χρηματοδοτικών προϊόντων. Δεν μάθαμε τα μαθήματα της κρίσης του 2009 εμείς. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε πλέον να υπαγορεύουν τους κανόνες κανόνες, μόνο οι αγορές. Η πολιτική είναι πάνω από τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον φιλοξενούμενό μας εκ ψενόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που τόσο πολλοί από εσά υποστηρίζετε αυτή την νομοθεσία η οποία θα αυξήσει την διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Κομισιόν θέλει να οριστικοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι κανόνες για την παροχή αναφορών. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε την γρήγορη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση των πυρηνικών κινδύνων και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή διαχείρισή του. Αυτή νομοθεσία ε, προβλέπει μέχρι το τέλος του 2016 να συνταχθεί μια έκθεση από την ΕΣΜΑ η οποία θα εξετάσει τις διάφορες προτάσεις. Η Κομισιόν θα δημοσιεύσει την έκθεσή της ένα χρόνο αργότερα και θα συζητήσει και για τις διεθνείς προσπάθειες που γίνονται για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές αξιογράφων. Αυτό θα περιλαμβάνει και τις προτάσεις του ε, <clears throat> Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αυτό όμως δεν εμποδίζει το να περάσουμε αυτή την νομοθεσία για να μειώσουμε τον κίνδυνο, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε να μπορούν οι επενδυτέ να κάνουν σωστέ επενδύσει και να γίνουν οι αγορέ μα πιο ασφαλεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν και ο, τώρα ο εισηγητής μας, ο κύριος Σόρου έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ε, θετικά αξιολογώ τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν σήμερα, σήμερα στην Ολομέλεια σχετικά με την θετική τους άποψη για το κείμενο το οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο. Ο Κλάφος Βάλλη μίλησε ε, τελευταίος και νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικά αυστηρός όπως και μερικοί άλλοι συνάδελφοι σχετικά με το ότι χάσαμε την ευκαιρία να βάλουμε ένα ε, όριο στο ε, δασμό που, τέλος το οποίο χρησιμοποιείται καθώς επίσης και τον αριθμό των, των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι τίτλοι. Έχουμε, μην το λησμονείτε, την Ευρωπαϊκή Αρχή ναι, για την παρακολούθηση των συστημικών ε, κινδύνων. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό λοιπόν ασχολείται με το θέμα ε, και νομίζω ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά και τους ελέγχους αυτούς και την παροχή της απαραίτητης ρευστότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω συναδέλφους και όδη συζητητές για την επικοδομητική τους συνεργασία καθώς και τους υπαλλήλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν ε, για την, ε, την ε, ΦΙΣΜ, καθώς επίσης και το Συμβούλιο, αλλά και την Ιταλική Προεδρία, η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, ειλικρινώς. Κύριε Σιγητά. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.